Right, good morning, ladies and gentlemen. Έχουμε, ο, προ... ο ήχος πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα, έτσι δεν είναι. Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Καλημέρα, αγαπητοί συναδέλφοι. Ακούστε και στο δωματίο είναι Ε, δεν είναι τόσο καλή, οπότε σας παρακαλώ εσείς τουλάχιστον να κάνετε ησυχία και να συνεχίσετε τις ε, κατεδίαν συζητήσεις εκτός εθούσης. Ε, κοινή συνεδρίαση ΑΦΕΤ ΑΦΚΟ βάσει του άρθρου 55 ε, σημείο 1 έγκριση πρακτικών της συνεδρίας 15 Δεκεμβρίου σχόλια όχι σημείο 2 έγκριση μέσης διάταξης σχόλια όχι. Σημείο 3. Συνταγματικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινή πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας που προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, θα διεξαχθεί η ψηφοφορία ε, στη, με τις δύο επιτροπές. Ε, κύριε Φλέκενσταν, ε, ναι, Προσπαθούσα το καλό να κάνω, αλλά τελικά την πάτησα. Εγώ αποσύρω τώρα την προφορική μου τροπολογία, ε, η 196. Πρέπει να το πω, μου είπανε πριν από την ψηφοφορία. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Φλεκενστάιν. Αποσύρεται 196 λοιπόν. Θέλω να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της ΑΦΚΟ. Σίλβα Περέιρα, εδώ είστε. Θέλετε μήπως να πείτε κάτι. Ευχαριστώ. Συγγνώμη για την αργοπορία. Σας καλωσορίζω. Το μόνο που θα ανέφερα είναι θα τόνιζα μάλλον είναι πόσο σημαντικό είναι το θέμα δεδομένου και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση και να αποφασίσουμε από κοινού για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ. Μα ευχαριστούμε τον Συμπρόεδρο εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς ε, τους εισηγητές και τις επιτροπές. Μίχελ Γκάλε, Έστεβαν κονσάλες Πόνς, οι συνεισηγητές μας, οι συνεισηγητές μας δεν θέλουν να πούνε κάτι. Αν συμφωνείτε λοιπόν να αρχίσουμε με την ψηφοφορία. Στις 10 παρατέταρτο θέλουμε να έχουμε τελειώσει. 35 λεπτά λοιπόν έχουμε στη διάθεσή μας για την ψηφοφορία. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και γρήγοροι. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα. Ε, τροπολογία 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ για την 147. Γιατί δεν δουλεύει το μηχάνημα. άρχισε η ψηφοφορία. ID error λέει εδώ. Αν έχω βάλει την σωστή κάρτα. 63 ψήφισαν, εγκρίθηκε. 148 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές, έλεγχος παρακαλώ, για τη συμβαστική εννέα. Closed. Πέρας. Σαφέστατα υπέρ ψηφίου. Συμβαστική ενέα εγκρίνεται και πάμε στις 170, 71, 72, 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 174 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτονται 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 178, 179 και 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 10 υπέρ Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Δεν είμαι σίγουρος. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίθηκε και φτάνουμε τώρα στις 189, 90, 91 και 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 193. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 196. Απεσύρθη. Άρα, ψηφίσουμε μόνο για το πρώτο τμήμα. Καλά τα λέω. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για το πρώτο τμήμα, της 196. Ψηφίζουμε για την 196, τμήμα 1. Χωρίς την προφορική τροπολογία, ευχαριστώ κύριε Φρακενστάν. Ευχαριστούμε για τις συμβουλές, αλλά ξέρουμε τι κάνουμε εδώ στο Προεδρείο. Είμαστε ενημερωμένοι. Μάλιστα, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 197, 198, 199, 200 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 203 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 204 υπέρ. Κατά. Αποχές. 205 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 206 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Και τώρα συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 232 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 233 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 234 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 236 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 237-238 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 239 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 240 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 241 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 242 υπέρ κατά αποχές Εγκρίθηκε. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 2.60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτω 2.61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Γιατί 2.61 ηλεκτρονική επαλήθευση. ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Τώρα γίναμε 68. Απορρίπτεται. 2,62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2,63 υπέρ. Συγγνώμη, τι ήταν, ένα λεπτό. καταπίτη, γιατί εγκρίθηκε η 2.32, 2.64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ε απορρίπτεται. 2.66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 269 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 270 υπέρ. Για τη 269 ζητάτε επαλήθευση. Πολύ καλά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Νομίζω ότι τώρα πιάνει ξεκάθαρα ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. 2,70 Λάινεν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2,71 υπέρ. Συγγνώμη, τίποτα. Κατά εδώ. Και άρα 2,73 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2,77 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2,78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2,79 και 2,80 υπέρ, κατά Αποχές. Απορρίπτονται. 281 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Γιατί 281. Άρχεται. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 282. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 283. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 284. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 285 και 286 που αποσύρθηκε και 287 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 288 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 289-290 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 291. Όχι. 289-290 ήταν σαφές το αποτέλεσμα, αλλά σε παληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Χαίρομαι ότι είμαστε ε, πλέον 70 παρόντες, λίγη ψηφοφορία, 58 κατά 12 υπέρ. Είναι σαφές. Ωραία. Πού είμαστε. 2.91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.92, 2.93, 2.94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 2.95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική υπαριθμό 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 303. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 304, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 305, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 306, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική Αριθμό 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 324. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Συμβαστική παριθμό 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Σαφής πλειοψηφία υπέρ. 338. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 339 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 340 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 341 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 342 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 343 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική παριθμό 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην 358 και 359 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 360 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 363 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 365 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική υπάρχουν 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 375 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 376 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 377 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 378 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 378. Ωραία, επαληθεύουμε την 378, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 39 υπέρ 30 κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην 379 του κ. Φανόρδεν Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 380. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 381. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 382, 383, 384 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 386 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 387 υπέρ. Κατά. Όχι, η 19, συμβαστική 19 υιοθετήθηκε, άρα αυτές οι δύο καταπίπτουν. Πού πάμε τώρα. Συγγνώμη, μια μικρή σύγχυση εδώ. Περνάμε στις 404 και 405. Καστάλτο κλπ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται, απορρίπτονται 406 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 407 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 408 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 409 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 410 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 411 υπέρ 410 υιοθετήθηκε, ωραία. Περνάμε στην 413. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 414 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 415 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 416 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 417 υπέρ όχι το 414 θετήθηκε όχι περνάμε λοιπόν στη συμβαστική υπαρθμόν 20 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται να επαληθεύσουμε όχι προφανές ε εντάξει Συμβαστική παραθμόν 20 εγκρίθηκε, άρα περνάμε στη συμβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτή εγκρίνεται. 436. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 437. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4.38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4.39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 440 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική παριθμόν 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 442 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 445 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 446 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 447 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 448 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 449 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.55 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 4.56 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 4.57 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμόν 23 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 458. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 στην αιτιολική έκθεση πλέον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Χωριστή ψηφοφορία που τη ζήτησε το ΕΛΚ. Τμήμα 1. Υπέρ. Κατά. Αποχής. Εγκρίνεται. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το επαληθεύουμε. Λίγη ψηφοφορία. 48 υπέρ 20 κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 24. Ο, οι συνεισηγητέ έχουν προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμών 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ. Κατά τα αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 και 73 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ. Ο άμε συγχωρείται. έκανα λάθος, καταπίπτει. 78 κατά συνέπεια του κυρίου Πιτίδιου υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 89 και 90 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. Η 18 ο έχει εγκριθεί νεάρα, ναι, η 92 καταπίπτει. 93. Όχι,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 99 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 100 και 102 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 101 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Εγκρίθηκε η συμβαστική 9. Ωραία. Τότε 110. Ψηφίζουμε την 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε καλύτερα 123 ελέγχουμε άρχεται η ψηφοφορία Δύο συνάδελφοι δεν συμμετέχουν. Εντάξει, κλείνει. Α, απορρίφθηκε μαζικά. 124 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 κατά, αποχές, ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε καλύτερα την 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έξι, παράγραφος 6, γνωμοδότηση υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Αν καταλαβαίνω καλά, έχουμε και μία τελική ψηφοφορία ως προς τη γνωμοδότηση, α, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά, ε, ως προς τη γνωμοδότηση όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Και η 70. Ωραία και να συγχαρούμε τον εισηγητή γιατί εγκρίθηκε αυτή η έκθεση. Τους εισηγητές μάλλον. Διαδικαστικό. Παρκ. Λέζιν. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της ΓΚΟΕ έχουμε συντάξει μία έκθεση μειοψηφία την οποία έχουμε αποστείλει και στη γραμματεία. Ευχαριστούμε για την πληροφόρηση αυτή. Ε, κάτι άλλο παρακαλώ. Κάποιος άλλος. Φαίνεται πως όχι. Τότε ευχαριστώ τους συναδέλφους της ΑΦΚΟ που παρευρέθηκαν και για τη συμμετοχή σας.